Κυρία Γκάμπριελ, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Όσο, όσοι θέλουν να βγουν, παρακαλώ να βγουν γρήγορα και ήσυχα. Περνάμε στις δηλώσεις ψήφου. Η πρώτη δήλωση, σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση, Ιζαμπέλ Τομά, για τον βορειοατλαντικό, βορειοανατολικό Ατλαντικό από θέματα βαθέων υδάτων και αλία σε διεθνή ύδατα. Ο κύριος Χάζεκαμπ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Σε λίγο πιάνουμε πάτο. Υπάρχουν 10 εκατομμύρια ζωικά και φυτικά είδη στους ωκεανούς μας. Πολλά